Ε, Καλή σας ημέρα, συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Το πρώτο θέμα της Μέσης Δάξεως είναι η δήλωση της Κομισιόν αφορικά με την τήρηση των εθνικών μισθολογικών συμβάσεων και των μηχανισμών συνταξιοδότησης. Έχουμε ανάμεσα στον Επιτροπογείο Χάννα, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλώς ορίσατε κύριε Χάν στο Κοινοβούλιο και στην σημερινή μα συζήτηση. Έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε την δήλωση της ε, Κομισιόν σχετικά με την ανακοίνωση. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη.